Ε, του Φράγκο από Συψεμία. Να δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφό μας ε, ε, Μέρ Κοστέλου. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ και τα μέλη και για το ενδιαφέρον που δείξατε για αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα για να καταδείξουμε την αλληλεγγύη μας με τους φτωχούς ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω το γεγονός ότι υπάρχει υποστήριξη για τα 3,5 δις και θα μας υποστηρίξει και το Συμβούλιο. Σε σχέση με τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα θα ήθελα να ε, διασαφηνίσω ορισμένα πράγματα, διότι ίσως οι λέξεις αυτές οδηγούν σε παρανόηση. Αυτό που έχει σημασία είναι τα προβλεπόμενα κονδύλια για τους απόρους να πάει να πάνε πραγματικά στους πλέον ενδέεις και η πρόταση που εγκρίναμε τον ε, προηγούμενο μήνα είναι ο τρόπος για να φτάσουμε σε αυτό. Υπάρχουν πολλά ε, θέματα σε σχέση με τις τροπολογίες των φιλελευθέρων και των πρασίνων και θα ήθελα να τονίσω ορισμένα ε, ζητήματα ως προς το περίπλοκο χαρακτήρα του συστήματος προειδοποίησης και εποπτείας. Μιλήσαμε για τον Ιανουάριο του 2014, γιατί μιλάμε για αυτή τη για αυτή την ευάλωτη κατηγορία ανθρώπων που ζουν στα περιθώρια, στο περιθώριο της κοινωνίας. Επίσης, δεν γίνεται επανακατανομή χρημάτων όπως προβλέπεται από τις τροπολογίες. Εάν το λύσουν ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το κάνουν μέσω του ΕΤΠΑ ή του ΕΚΤ. Θα ήθελα επίσης να πω ότι οι οργανώσεις των κρατών που δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα ε, διατροφ, διατροφικών αναγκών θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι αν υπάρξει αλλαγή σε κυβερνητική πολιτική η αλλαγή κυβέρνησης, τότε τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, όπως είπε και η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, γιατί αυτά τα χρήματα είναι για ανθρώπους, όχι για κυβερνήσει, που ζουν σε, κατάσταση απόλυτης ένδυας. Ελπίζω να μας επιτρέψει ψέτε να φτάσουμε στους στόχους του 2020, να μειώσουμε δηλαδή τον αριθμό των εμβεών κατά 20 εκατομμύρια. Ευχαριστούμε, Έμερ. Κλείνει η συζήτηση, η οποία ήταν ιδιαίτερα ζωηρή με πολλαπλές παρεμβάσεις. Νομίζω ότι είναι μία από τις συζητήσεις που μας δίνουν, ενισχύουν την αξιοπιστία μας και η ψηφοφορία θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Ε, τώρα, αλλά το θέμα αυτό θα ψηφιστεί αύριο στις 11.30. Ε, τώρα θα περάσουμε στην ώρα των ψηφοφοριών που θα αρχίσουν σε 2-3 λεπτά. Διακόπτουμε λοιπόν για 2-3 λεπτά μέχρι ότου καθίσετε όλοι και ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση χωρίς να ε, ανακύψουν, χωρίς να υπάρξει, να με ησυχία εν πάση περιπτώσει και χωρίς να ανακύψουν επεισόδια.